Ε, Αγαπητοί φίλοι, έχουμε πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε, έχουμε μια τόσο σημαντική ακρόαση και ορισμένοι συνάδελφοι με ενημέρωσαν πριν από μισή ώρα, πριν από μία ώρα, ότι έπρεπε να φύγουν, να πάνε στο αεροδρόμιο. Γιατί πρέπει να πάνε δυόμιση και τρεις ώρες πριν την πτήση τους. Άρα δεν έχουμε συναδέλφους βουλευτές παρόντες. Και από την άλλη όμως, είμαι και σε πολύ δεινή κατάσταση. Γιατί εγώ πρέπει να φύγω στις 4. Και μέχρι τις 5.30 έχουμε προβλέψει την ακρόαση. Οπότε για μένα δεν θα ήταν πρόβλημα. Από την άλλη λέει ο κύριος Έριξον, είναι παρόντες ε, και άνθρωποι που είναι σημαντικοί οι ίδιοι. Οι παρόντες έχουν σημασία. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά, λέει ο πρόεδρος, ακούω φωνές. Α, ο κύριος Έριξον. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ λογικό αυτό που είπατε και πάρα πολύ εύστοχο, κύριε Έριξον, και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας είναι. Τι προτείνω τώρα εγώ. Να προχωρήσουμε, να ακούσουμε το πρώτο πάνελ. Μάλλον να, κάνουμε τα δύο πάνελ ένα, να μιλήσουν όλοι οι ομιλητές. 7-8 λεπτά παρακαλώ έκαστος, αν γίνεται. Και μετά να γίνει συζήτηση και μεταξύ σας το μελών του πάνελ, γιατί έτσι θα συγχωνεύσουμε τα δύο πάνελ σε ένα και ε, μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις στα μέλη των δύο πάνελ που μπορεί να μην έχουν πάντα τις ίδιες ε, θέσεις, απόψεις ε, και να τελειώσουμε νωρίτερα, μισή ώρα, 40 λεπτά νωρίτερα, κάτι τέτοιο. Συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Ε, ναι, να περάσουμε αμέσω στην ουσία δεν σας ρωτώ καν αν συμφωνείτε. Βλέπω ότι συμφωνείτε και προχωρώ. Mm. Uh, λοιπόν, βλέπετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Συνήθως ε, στην αρχή κάνω μια σύντομη παρουσίαση 5-7 λεπτά. Δύο-τρεις προτάσεις μόνο ο ρόλο τη αποθήκευση ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μελλοντικό σύστημα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα και για το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, αυτό που ε, είναι το θέμα είναι η αποθήκευση. Η ε, ΑΠΕ, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και πάλι η αποθήκευση. Όλα τα θέματα ουσία εκεί βρίσκονται. Μπαίνουμε λοιπόν κατευθείαν στην ουσία και θα δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή μα, που είναι ο κύριος Πατρίκ Κλέρεν, γενικό γραμματέα. Ε, ε, της ε, Ένωσης για την Αποθήκευση Ενέργειας. Συνήθως παρουσιάζω και συστήνω τα μέλη του πάνελ, αλλά νομίζω ότι και αυτή τη φορά μπορούμε να συντομεύσουμε και να... Έτσι κι αλλιώς σας γνωρίζουμε πάνω κάτω, πολλοί από εμά δεν είστε άγνωστοι. Παρακαλώ κύριε Κλέρενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αρχισογραφίας, ονομάζομαι Πατρικλάνη, είμαι γενικό ε, γραμματέα του ΕΑΣ, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αποθήκευση ενέργεια. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο. Έχουν περάσει ήδη 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο ΙΖ λοιπόν, έχει τρει βασικού ε, σκοπού. Πρώτον, να διαμεράσουμε σε εσά και άλλου το όφελο τη αποθήκευση ενέργεια να έχουμε έναν ε, κατάλληλο και δίκαιο ε, μηχανισμό στην αγορά και σχεδιασμό της αγοράς και να προωθήσουμε την ε, αποθήκευση ενέργειας για να έχουμε χρηματοδότηση για την έρευνα και την προβολή των τεχνολογιών. Και θα δείτε ότι τα μέλη μας είναι πολύ άριθμα, περίπου 40. Εκπροσωπούν και τα ερευνητικά κέντρα, τους παρόχους εξοπλισμού, τις εγκαταστάσεις, τους TSOs. όλες συμμετέχουν. Αφενός λοιπόν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, έχουμε την πρόκληση γιατί όλοι πρέπει να μιλούμε με, μια φωνή, ακόμα και ανταγωνιστές και από την άλλη ο ΙΖ εκπροσωπεί το σύνολο του κλάδου και όχι μόνο ένα ή άλλο τμήμα του. Ήθελα σήμερα να σας δείξω ότι στο πλαίσιο της αποθήκευσης ενέργειας έχουμε επιμέρους τεχνολογίες. Δεν είναι μία και μοναδική. Γι' αυτό και είναι τόσο περίπλοκη η κατάσταση. Έχουμε πέντε. Την, την χημική, ηλεκτρική, ηλεκτροχημική, μηχανική και θερμική μορφή αποθήκευσης ενέργειας. Ουσιαστικά τα μέλη των οικογενειών αλλάζουν, αλλά οι οικογένειες παραμένουν περίπου ίδιες. Θα δείτε λοιπόν στη συνέχεια ότι έχουμε και το υδρογόνο και συνθετικά δίκτυα φυσικού αερίου. Έχουμε διάφορες ε, μορφές ε, με μηχανικές ε, αντλίες και την αποθήκευση. Όλα αυτά έχουν προσθεμένη αξία και όλα συμβάλλουν για την εξορρόπηση του συνολικού συστήματος. Θα δείτε η επόμενη διαφάνεια είναι εξαιρετικά τεχνική. Θα δείτε ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι παντού και στις κατοικίες και στη βιομηχανία. Μπορούμε να διευκολύνουμε την παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και την αιωλική, διαδραματίζει ρόλο παντού. Γι' αυτό και έχουμε επιμέρους διαφορετικές τεχνολογίες με διαφορετικές υπηρεσίες που ε, συνεισφέρουν ε, στο συνολικό σύστημα. Γι' αυτό απαιτείται και αυτή, ε, αυτές οι ιδιαιτερότητες απαιτούνται. Προσπαθούμε να σας δείξουμε ότι υπάρχει στήριξη από την παραγωγή στη συμβατική αλλά και στις νέες μορφές δεν θα τα διατρέξω όλα. Έχουμε και το σύστημα μετάδοσης, μεταφοράς και πολύ συχνά είναι πολύ ταχύτερη αυτή η οδός. Για παράδειγμα, ε, σε ένα μιλισεκόντ μπορεί να ξεκινήσει κανείς μια μπαταρία, έχει δηλαδή διαθέσιμη την ενέργεια. Αν θέλει ε, κανείς να ξεκινήσει ένα ε, μια άλλη διαφορετική εγκατάσταση παραγωγής, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Επομένω, αυτό βοηθάει και τον καταναλωτή. Και αυτό θα θέλαμε να δείξουμε, ότι δεν υπάρχει μία και μόνη τεχνολογία που είναι η ιδανική. Είναι ένα μείγμα διαφορετικών τεχνολογιών. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα επιμέρου στοιχεία. Και αυτέ τι τεχνολογίε θα εξελιχθούν. Επομένω, όταν αποφασίσετε ένα νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο που οι τεχνολογίε να, να έχουν δυνατότητα να εξελιχθούν και να μην ε, τι ε, παρεμποδίζετε. Να είναι ανοιχτό και με δυνατότητε προσαρμογή, λοιπόν, το καθεστώ. Είχαμε ακρόαση και με τις πολιτικές ομάδες και εκεί δώσαμε και κάποια παραδείγματα. Ε, σε επίπεδο διανομής έχουμε πολλές ε, ε, μορφές, ε, ιδίως σε ό,τι αφορά το επίπεδο ε, φωτοβολταϊκών και θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Ε, έχουμε ζητήματα ποιότητας, από πλευράς ανταπόκριση στη ζήτηση. αν έχει κάποιος μια, ένα σωρευτή θα μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει αν θα το συνδέσει με το δίκτυο ή όχι, ανάλογα με το χρόνο που είναι φθηνότερη η ηλεκτρική ενέργεια και μετά να το οικοδομήσουμε από εκεί και πέρα. Δεν χρειάζεται κάποιο να φτιάξει με τεράστια εγκατάσταση, να βάλει κάποια πέτρη πλάξη και μετά να προσθέσει. Αλλά και από πλευρά TSO ε, υπάρχει ευρύτατη στήριξη. Δεν θέλω να τα αναφέρω όλα αναλυτικά, όμω αυτό επιτρέπει την ταχύτατη εξισορρόπηση του συστήματο. Και μετά για τους παραγωγούς καταναλωτές, prosumer, κάτι το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε όλοι, θέλουμε ε, να δώσουμε αυτές τις δυνατότητες και στους καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν και αυτή την ε, πλευρά από την αποθήκευση ε, θερμικής ενέργειας, ε, σωρευτών, πολλές μορφές αποθήκευσης ενέργειας υπάρχουν και δεν είναι απαραίτητα πιο φθηνή ηλεκτρική, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μπορεί εδώ να είναι πιο φθηνή ορισμένες φορές. Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός αγοράς στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται ε, στην ιστορική εξέλιξη. Επομένως, κατά κύριο λόγο εξετάζει την κεντροποιημένη παραγωγή ενέργειας. Και προκειμένου να έχουμε ολόκληρο το, το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο, πρέπει ε, να ενσωματώσουμε εκεί και την παραγωγή ενέργειας. Και το θέμα είναι ποιος ε, είναι ιδιοκτήτης. Είναι βάσει των ε, προσπαθειών παραγωγής ή δεν είναι περισσότερο στοιχείο παραγωγής, επομένως μπορεί να είναι και καταναλωτής μια εγκατάσταση αποθήκευση. Γι' αυτό έχουμε και μια τέταρτη κατηγορία, τέταρτο στοιχείο του ενεργειακού συστήματο. Και μετά βλέπουμε ότι η εφαρμογή αυτή τη ε, αποθήκευση ενέργεια ορισμένε φορέ είναι δύσκολη ε, εξαιτία των συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Φόροι, τέλη. Ε, είναι διπλή φορολόγηση, χωρίς κάποιος να καταναλώνει την ενέργεια πρέπει να, να υπάρχει αυτή η διπλή φορολόγηση και για τη φόρτωση και για την ε, απελευθέρωση. Μετά, οι ανανεώσιμε. ανανεώσιμες. Ξέρετε ότι με τις ε, dispatchable μορφές θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ, μορφές θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ ε, περισσότερη ευελιξία στο σύστημα. Όλες οι υπηρεσίες αγοράς ε, υπηρεσίε ε, των συστημάτων θα πρέπει να υπάρχουν στην αγορά. Κανένα παραγωγό δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παράσχει μια υπηρεσία. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, αν κάποιο ω παραγωγό δεν μπορεί να πουλήσει όλη του την ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να διατηρήσει ένα τμήμα του για τον TSO. Και λέμε ότι δεν είναι δίκαιο να του ε, υποχρεώνουμε, να τα τεθούν όλα αυτά στην αγορά και η καλύτερη τιμή θα υπερισχύσει. Επίσης, αν δώσει κάποιος καλύτερη υπηρεσία στο σύστημα, δεν έχει καλύτερη ανταμοιβή. Δεν θα πάρει κάποιος περισσότερα χρήματα. Άλλοι θα πάρουν την προστιθέμενη αξία, αλλά δεν θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Να πληρώνουμε βάση ε, των επιδόσεων. Και χρειαζόμαστε ασφάλεια με τις νέες ε, τεχνολογίες, δεν θέλουμε ε, άλλη στήριξη, αλλά να υπάρχουν μακροπρόθεσμες συμβάσει προκειμένου να μπορεί κανεί να επενδύσει ε, και να υπάρξει και απόσβεση. Για να μπορεί ας να έχει ένα ε, οκταετές, πλαίσιο και να μπορεί να πάει στην τράπεζα. Αυτό εν συντομία. Πολλέ τεχνολογίες με προστιθέμενη αξία, με διαφορετικέ μορφέ. Θα πρέπει να προσαρμοστεί ο ε, κλάδος της αγοράς, ο σχεδιασμό της αγοράς και δεν ζητούμε οικονομική στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Είστε εξαιρετικά γνωστό, ε, κύριε Κλέρενς, γιατί αλλάξατε εκ βάθρων την ε, κατάσταση σε ό,τι αφορά ε, την ένωση αυτή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια γιατί από 13 μέλη το 2011 πήγατε στα 40. Τριπλασιάστηκαν λοιπόν τα μέλη σα. Και ασχολείστε και με τα ζητήματα τα κλιματικά και τα ενεργειακά το 2003. Επομένω, ε, κάποιοι από εμά ε, σα γνωρίζουμε από παλιά εδώ στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στόχος Χαμαχερέ έχει το λόγο τώρα έχει σπουδάσει φυσική σε πολλά μέρη. Ίσως δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο κύριος Κλέρενς, όμως ε, στη Βόνη, στο Άχεν, στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια, αλλά και στο Ινστιτούτο Μαξ Φλάνκ. Είστε μέλος ε, του Κέντρου Περιβαλλοντικών Επιστημών ε, του Πανεπιστημίου του Αυσβουργού. Παρακαλώ. Ο Augsburg. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Ε, θα σας δώσω θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γενική έποψη για το πώς ε, βλέπουμε ε, αυτό το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Το βασικό ερώτημα που κρύβεται είναι πώς μπορούμε να εντάξουμε τις απέτησες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι το βασικό πεδίο στο οποίο εργαζόμαστε. Και εξετάζοντας αυτά, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε ε, αυτό το θέμα, να δούμε ποιες είναι ανταγωνιστικές τεχνολογίες και πώς αλλιώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, σας έχω εδώ τέσσερα σημεία που θεωρώ πιο σημαντικά να εξετάσουμε όταν προσπαθούμε να ε, συγκρίνουμε τις άλλες δυνατότητες. Το ένα είναι ότι μπορεί να έχουμε μεγάλα δίκτυα και θα πω δύο λόγια. Μια που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ευρωπαϊκό εγχείρημα οι ανανεώσιμες από όλη την Ευρώπη ε, να συγκεντρωθούν με τη διαφοροποίησή τους και τη διαφοροποίηση αυτή να την κάνουμε ισχύ μας. Ε, επίσης η ε, ζήτηση είναι ελαστική. Στο μέλλον θα έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούν να ε, φορτίζουν ε, όχι μόνο όταν είναι στην πρίζα, ε, αλλά να μπαίνουν και στην πρίζα όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνδέονται διάφοροι τομείς. Δηλαδή, ένα σύστημα ηλεκτρισμού να συνδέεται με ένα σύστημα θέρμανσης και είναι τεράστιες αυτές οι δυνατότητες που διανοίγονται για τις επόμενες δεκαετίες για να απορροφηθούν όλες οι διακοιμάνσεις και να μπουν ε, και στη θέρμαση ανανεώσιμες, δηλαδή με ένα σβάρο δυο τριγών. Και μετά έχουμε και το θέμα της αποθήκευσης ε, του ηλεκτρισμού. Έχω πάρα πολλές διαφάνειες, υπερβολικό αριθμό. Το μόνο που θέλω να σας δείξω είναι το εξή. Κοιτάξτε τι γίνεται με την νεολική ενέργεια, από χώρα σε χώρο, πώς διαφέρει έχουμε ε, αυτή την διακύμαση, δεν θα το εξηγήσω σε λεπτομέρειες, αυτή την καμπύλη. Αν δείτε την Ευρώπη, το κόκκινο, το, το πράσινο είναι η Γερμανία και το μπλε είναι μία συγκεκριμένη χώρα άλλη. Όταν δημιουργούμε μεγάλα δίκτυα, ε, απορροφάται η αιωλική ενέργεια και μειώνεται και η ανάγκη για αποθήκευση. Η Ευρώπη ε, είναι παγκοσμίω ε, από τις μεγαλύτερες περιοχές που έχουν αρκετό αέρα. Μόνο στη Βόρεια Θάλασσα σκεφτείτε πόσο φυσάει ο άνεμος. Έρχομαι τώρα στην αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας και βλέπω την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Έχω μερικές διαφάνειες και φωτογραφίες από τη Γερμανία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αρκεί να δει κανείς το ηλεκτρικό σύστημα ε, και τους, ε, τα ποσοστά δίζησης των ΑΠΕ για να φτάσουμε στο 80% για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε αποθήκευση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποθηκεύεις μόνο ως συσσωρευτή ε, καλύπτει τις ανάγκες της ε, ε, μέρας, τη νύχτα και αντίστροφα, αλλά ε, πρέπει να καλύπτουμε και τις διάφορες εποχές του χρόνου. Και κάθε φορά που χρειάζεται τέτοια εξισορρόπηση, χρειάζεται υδρογόνο. Κάτι πολύ περίπλοκο από το να έχεις, ξέρω εγώ, στο υπόγειό σου μια μπαταρία να Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και από όλα αυτά που σας δείχνω από τις τόσες πολλές διαφάνειες τις οποίες διατρέχω είναι ότι αυτό θα έρθει αργά χρονικά όταν φτάσουμε σε πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων στο μείγμα μας και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αν το δούμε έτσι χρειάζεται λιγότερη αποθήκευση ή μόνο σε εθνικό. Και έρχομαι τώρα στην ε, σύνδεση των διαφόρων τομέων sector coupling, που είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τους διάφορους κλάδους. Όταν φέρνεις ηλεκτρική ενέργεια μέσα σε ένα σύστημα θέρμανσης, αυτό μπορεί να έχει πολλές ευεργετικές συνέπειες. Μπορούμε να έχουμε μεγάλες αντλίες που θα παίρνουν την ηλεκτρική ενέργεια και να ε, την πολλαπλασιάζουν, να την τριπλασιάζουν κτλ. Ε, μπορούμε λοιπόν να φέρουμε ε, στο boiler ε, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες. Μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει κάποια αδράνεια και μπορούμε να έχουμε και μια ελαφρά αποθήκευση της θερμότητας. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία βέβαια, χάνουμε σε αποτελεσματικότητα. Όταν έχουμε λοιπόν ηλεκτρική θέρμανση στη θέρμανση μιας ολόκληρης περιοχής, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγάλες ε, ε, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 10 με 15 κιλοβατόρες ας πούμε Μάλλον, μάλλον 10 με 15 ευρώ ανά κιλοβατόρα, διορθώνει ο μιλητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν και θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το δρόμο. και βλέπουμε τώρα την αποθήκευση μέρα, νύχτα, εβδομαδιαία, ε, ένα σύστημα θέρμανσης ολόκληρων περιοχών και πώς αυτό μπορεί να διευκολύνει ε, την ε, διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αν έχουμε ένα σύστημα λοιπόν σύνδεσης με αποθήκευση, δεν αποθηκεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αποθηκεύουμε τη θερμότητα. Ένα σύστημα που βασίζεται μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται τεράστια εγκατάσταση υδρογόνο κτλ. Ε, αν καταφέρουμε λοιπόν να συνδέσουμε τη θέρμανση με το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λοιπά και να δημιουργηθεί τέτοια δυνατότητα στην αγορά, τότε φυσικά αλλάζουν τα πράγματα και ε, Ξέρετε ότι υπάρχει σήμερα η τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολλά από τα πράγματα αυτά ε, είναι στο στάδιο της ε, επίδειξης και μπορούν να μεταφραστούν και στην πράξη. Άρα λοιπόν και έρχομαι ήδη στην σύνοψή μου για να κλείσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε ε, την παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη. Έχουμε ηλιόλουστες περιοχές στο νότο, περιοχές με πολλούς ανέμους στο βορρά. Εγώ πολιτικός δεν είμαι βέβαια, αλλά θα μπορούσε αυτό να είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο. Κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι να το προωθήσουν και θα μας βοηθούσε. Το δεύτερο. Βεβαίω χρειαζόμαστε συστήματα αποθήκευσης, αλλά δεν έχω ε, Προκαταλήψει για το ποια τεχνολογία θα επιλέξουμε. Υπάρχουν διάφορε δυνατότητε και πρέπει να το αφήσουμε ανοιχτό. Και η σύνδεση των διαφόρων συστημάτων είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη έρευνα και ξέρω πάντα το λένε αυτό οι πανεπιστημιακοί μάλλον, αλλά χρειαζόμαστε ένα αυστηρό ε, κανονιστικό πλαίσιο και σε επίπεδο διανομής να φέρνει στην αγορά ανταγωνισμό. Είτε αποθήκευση είτε σύνδεση διαφόρων μορφών θα δούμε. Ε, και τέλος να πω κάτι ερετικό ίσως και προκλητικό, να σκεφτούμε και το θέμα εάν όλα αυτά που κάνουμε αυτές τις μέρες ε, είναι κάτι που συνάδει με την απελευθέρωση της αγοράς. Θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο πάρα πολύ ελεύθερο και απελευθερωμένο στην ηλεκτρική ενέργεια αν είχαμε πλήρη απελευθέρωση, θα να λειτουργούσαν καλά, αλλά και τα παλιωμοδίτικα, πιο κρατικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι άσχημο. Ξέρω ότι πολλούς ε, δεν τους ικανοποιεί αυτό. Η Ευρώπη λειτουργούσε πολύ καλά ε, με μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα έχουμε περάσει στην απελευθέρωση. Δεν είναι πάντα κάτι το θετικό. Σας είπα, αιρετική είναι αυτή η παρατήρηση. Και τέλος, ένα τελευταίο. Είναι σημαντικό στην πολιτική συζήτηση. Τα φωτοβολταϊκά και οι συσσωρευτές ε, θα πρέπει να συνδυαστούν παντού στην Ευρώπη και στην Αφρική, αν δείτε σε πολύ μικρά αφρικανικά χωριά τι μπορεί να φέρει ε, ένα σύστημα φωτοβολταϊκών μαζί με σωρευτές μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ω συνήθω οι καθηγητέ μακρηγορούν, αλλά έχω και εγώ αυτή την αδυναμία και τη μοιράζομαι μαζί σα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ καθηγητά και προχωρούμε στον επόμενο μιλητή. Έχω το προνόμιο να σας συστήσω και να καλωσορίσω φυσικά το Γιώργο Χατζημαρκάκη, πρώην Ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής Ήτρε για δύο θητείες, αν θυμάμαι καλά. Δέκα χρόνια. Πάρα πολύ δραστήριο μέλος στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, τη σχετική προετοιμασία και ήταν από τους πιο υπέρμαχους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και ε, Τεχνολογίας. Δεν ήμασταν πάρα πολλοί, 5-7 βουλευτές αγωνιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος Μπαρόσο. Ήταν πάντα πολύ ευγενή απέναντί μα. Λοιπόν, ο κύριο Χατζημαρκάκη τώρα είναι Γενικό Γραμματέα του Hydrogen Europe. Είχε και άλλε ιδιότητε τα τελευταία χρόνια. Αφού του ε, έφυγε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει σπουδάσει σε πολλά πανεπιστήμια και είναι πολύ γνωστός και μη εξαιρεταίος ο κύριος Χατζημαρκάκης. Και είναι και τα γενέθλιά του. Thank you very much. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γέρζη κύριε Πρόεδρε, που με καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Εγώ θα βουτήξω στα βαθιά κατευθείαν, γιατί περιμένω και τη συζήτηση. Η Hydrogen Europe, όπως βλέπετε εδώ, είναι μια ένωση 94 εταιριών από 16 κράτη-μέλη. Πρόκειται για μεγάλες εταιρείες όπως η Diamond, Siemens, Air Liquid, Linde, ε, και πολλές μικρομεσαίες. 50-50 είναι δηλαδή γιατί μας καλέσατε τώρα. Νομίζω ότι εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε πώς το υδρογόνο συγκρένεται με άλλες τεχνολογίες ε, αποθήκευσης είναι αέριο, αλλά επειδή μπορούμε μέσω της ηλεκτρόλυσης που είναι απλός τρόπος να το φτιάξουμε, ο ηλεκτρισμός ε, χρησιμοποιείται για να χωριστεί το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο και το αντίστροφο γίνεται πάλι, μπορεί πάλι να δημιουργηθεί ε, ηλεκτρισμός και άρα χρησιμοποιείται σε ένα εξαιρετικό ενεργειακό νέκταρ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, αμφίδρομα. Λοιπόν, ε, λόγω αυτής της ευελιξίας του ε, το υδρογόνο χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλους όγκους, το βλέπετε και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια. Ε, είναι βραχυ, βραχυπρόθεσμα. Οι εγκαταστάσεις για ηλεκτρόλυση χρειάζονται επενδύσεις. Βλέπετε ένα, μοντέλο εδώ στην είσοδο, αλλά είναι μεγάλο το κόστος, όμως η χρήση του υδρογόνου είναι ένας πολύτιμος ε, τρόπος για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Εδώ θέλω να σας δείξω ένα σύντομο ένα σύντομο βίντεο, βέβαια δεν παίζει τώρα εδώ, είναι πραγματικά 50 δευτερόλεπτα. Μπείτε στο Coloroid, ε, δείτε Coloroid υδρογόνο στην Google και γιατί χρησιμοποίησαν αυτό. Νικόλ Ρόιντ έχει, είναι ένας ε, λιανοπολιτής, ο μεγαλύτερος Βέλγος με 200, εταιρεία, με 200 καταστήματα στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε πράσινη ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα. Ο κύριος Κολρόιντ είναι δισεκατομμυρίουχος και αυτές ε, τα κλάρκα δεν λειτουργούσαν έπρεπε να τα φορτίζει όλη την ώρα. Ε, γι' αυτό έχει τώρα εγκαταστήσει στα δυτικά της των Βρυξελών, πολύ κοντά στις Βρυξέλλες, ε, ε, ε ανεμογεννήτριες και σε αυτό σε με κοινή κοινοπραξία με την χρήση υδρογόνου. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, ξέρω ότι ενδιαφέρεστε να τα δείτε και εσύ και ο Γεύζη και ο Πάουλ. Ε, δουλεύει τέλεια το σύστημα τώρα. Εδώ για να συνοψίσω να σας δείξω ότι το υδρογόνο είναι ένας διευκολυντής. Από τη μια έχουμε τη ε, δημιουργία ενέργειας πράσινης, ε, το ιδανικό, ηλιακή κτλ. Μετά το υδρογόνο αποθηκεύει μέσα σε αγωγούς, δεξαμενές ή ό,τι θέλετε και αργότερα μπορεί να γίνει εφαρμογή μέσω ε, μέσω, καύ, μέσω καύσης και όχι μόνο για διάφορες χρήσεις. Ε, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε το παράδειγμα ενός από, μιας από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης στην Ευρώπη. Είναι το πάρκο, ενεργειακό πάρκο του Mainz, Siemens, Lieben και Mainz Urban Utilities. Επίσης θα δείτε στην είσοδο ένα, μια μακέτα. 6 μεγαβατόρες ε, παράγονται για το πλέγμα, το grid. μετατρέπει την ενέργεια σε υδρογόνο που αποθηκεύεται σε, αυτά τα, σε αυτές τις δεξαμενές που βλέπετε που μοιάζουν με βιτία. Και μετά διοχετεύονται στις, ε, στους αγωγούς. Τι μπορεί να κάνει κανείς με το υδρογόνο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για και την κινητικότητα. Όπως βλέπετε για τα τρία αυτοκίνητα, τα επιβατικά ε, αυτοκίνητα που είναι στην, ήδη στην αγορά, το Hyundai X35, το Yota Mirai Αυτά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά από τον περισμένο Σεπτέμβριο και βλέπετε και ε, το Daimler B-Class στο μέσο. Βλέπετε και μικρά επαγγελματικά φορτηγά και λεωφορεία, αλλά και Clark. Ε, τα λεωφορεία κυκλοφορούν σε πάρα πολλές χώρες, έχουν φτάσει σε οριμότητα στις αγοράς, όπως και τα αυτοκίνητα και έχουμε και εδώ και ένα ωραίο ποδήλατο εδώ μπροστά μου. Πολύ ωραίο σχέδιο και με 60 γραμμάρια υδρογόνου μπορείς να τρέξεις 100 χιλιόμετρα με αυτό το ποδήλατο. Πολύ μεγάλη εμβέλεια δηλαδή. Και εδώ βλέπετε μια σύγκριση της εμβέλειας. Τι μπορεί κανείς να κάνει με το υδρογόνο. Αν συγκρίνουμε το κανονικό, την κανονική βενζίνη, ε, σε 4 λεπτά σου δίνει 500 χιλιόμετρα, ενώ το υδρογόνο θέλει λιγότερο από 5 λεπτά για να σου δώσει 500 χιλιόμετρα πάλι. Και τώρα, για να φορτίσει μια μπαταρία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε πάρει το γρηγορότερο φορτιστή Τέσλα που είναι 7 λεπτά για 20 ε, ε, λεπτά συγγνώμη, για 160 χιλιόμετρα. Ε, Βλέπετε ότι το υδρογόνο είναι ο μόνος τρόπος για να στραφούμε στον ηλεκτρισμό, στην κινητικότητα, χωρίς να αλλάξουμε τις συνήθειέ μα, γιατί μπορεί να τον γεμίσεις χωρίς πρόβλημα. Αύριο εγκαινιάζεται ο πρώτος ε, δωρεάν σταθμός ε, ανεφοδιασμού στο Βέλγιο, εδώ στο Ζάβεντεμ. Ξέρω ότι εσείς δεν θα είστε, αλλά οι βοηθοί σας θα έρθουν ένα λεωφορείο υδρογόνου, θα φύγει αύριο στις 12.30 από το Κοινοβούλιο και θα πάει όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σταθμό θα είναι και πολλά αυτοκίνητα υδρογόνου και όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο μπορεί να το καβαλήσει και να πάει. Αλλά ε, υπάρχουν δυνατότητες και άλλες για τη χρήση του υδρογόνου, για την θέρμανση, για την ψήξη. Εδώ έχουμε ένα κέντρο στοιχείων. Η Google είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής, αγοραστής μάλλον, πράσινης ενέργειας στον κόσμο. Δεν το ξέρω και εμένα με εξέπληξε αυτό. Όμως το πρόβλημά τους είναι τα κέντρα δεδομένων. Και τι κάνουν, το backup γίνεται μέσω του πετρελαίου γιατί είναι το πιο αξιόπιστο. Με, με κάλεσαν για να παρουσιάσω το υδρογόνο και τους άρεσε πάρα πολύ, διότι τους δίνει ενέργεια ασφάλεια ανεφοδιασμού και είναι και καθαρή ενέργεια, πράσινη ενέργεια. Και πιθανά θα αλλάξουν λοιπόν. Αν γίνει αυτό πραγματικότητα στην Ευρώπη σχεδόν, αλλά θα δείτε στην Ιαπωνία, η Ιαπωνική κυβέρνηση αποφάσισε να ονομάσει τους Ολυμπιακούς του 2020 του, του Τόκιου ε, τους αγώνες του υδρογόνου. Μετά το Φουκουσίμα ε, θα βάλουν νέες, νέα μηχανήματα για τη χρήση του υδρογόνου. Το έχουν αποφασίσει και λειτουργεί. Γιατί δεν υπάρχει όμως αγορά για την αποθήκευση. Αυτή είναι μια ερώτηση που έθεσαν οι προηγούμενοι μιλητέ. Εγώ σας έφερα μια μελέτη που έχει εκπονηθεί από την κοινοπραξία χρήση ε, καυσίμων και υδρογόνου. Θα την βρείτε τη μελέτη εδώ, στην είσοδο. Δεν υπάρχει αγορά ακόμα, δεν υπάρχει ορισμός και αυτό είναι ένα θέμα για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχουν κίνητρα για αποθήκευση. Ο κύριος Κόκλης ε, χαμογελά γιατί το λέει εδώ και πολλά χρόνια, το ξέρω. Και η ανεπάρκεια παραγωγής πλεονασμάτων, χωρίς να τα βάλει δηλαδή κανείς ε, στο grid, στο πλέγμα, δεν, δεν μπορείτε να το φανταστήσω. Πέρυσι χάσαμε ένα δις. Ένα δις. Γιατί δεν εφαρμόζεται ακόμα. Ε, αυτό είναι το θέμα της κότας και του αυγού. Υπάρχουν διάφορες ρυθμιστικές προκλήσεις. Χρειάζεται ξεκίνημα μιας αγοράς ανανεώσιμου υδρογόνου Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη. Κάποια υπάρχει, αλλά όχι αρκετή. Κίνητρα πρέπει να σχεδιαστούν για να αυξηθεί η ευελιξία του συστήμα, των συστημάτων ηλεκτρισμού. Ο κ. Κόχλη το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά και τι εννοώ ακριβώ. Εξαιρέσει ε, για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας από τον ε, Στη φορολογία του τελικού χρήστη δεν γίνεται και δεν, και δεν είναι επαρκή η αναγνώριση του υδρογόνου ως ε, πράσινου καυσίμου. Τι σου είπα Γιάννη, αν πάμε εδώ από το 0 μέχρι το 14 με τον ανελκυστήρα εδώ του Κοινοβουλίου θα σας πω ότι το υδρογόνο είναι το πιο ευέλικτο στην αποθήκευση ε, επίσης είναι ο, η, κρίκος που λείπει στην αλυσίδα για να, να καταργηθεί η χρήση του άνθρακα μέχρι το 2050. Επίσης ε, είναι το μόνο καύσιμο που επιτρέπει ε, την ίδια κινητικότητα χωρίς αλλαγή συνηθιών και έχει και τα μεγαλύτερα ψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ πως και οι πολιτικοί μακρηγορούν ελαφρώς περισσότερο από τους καθηγητές. Ε, ναι, αποκάλυψη για μένα. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν όλοι ξέρετε ο Ευχαριστώ Γιώργο. Βλέπουμε ότι έχει πάθο ε, σε όσα κάνει. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Μπεν Χιλ, που είναι αντιπρόεδρο τη Tesla Energy. Ε, αναφέρατε την Tesla στην ομιλία σα. Ο κύριο Μπεν Χιλ ασχολείται με την ηλεκτρονική, με την ηλιακή, τον ηλιακό ηλεκτρισμό από το 1986, πολύ καιρό. Και τώρα ηγείται των φιλοδόξων δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων της Τέσλα στην Ευρώπη και στην Αφρική. Εμπορικές και ενεργειακές ε, δράσεις, δραστηριότητες και στην Αφρική για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ενδιαφερόμαστε πολύ να σα ακούσουμε και να σα πω, συνάδελφοι, γιατί είναι αυτό και στο πρόγραμμά μα. Πρώτα έχουμε δύο ομιλίε, ενώ με τους κύριους μας ε, ε, το κύριο μας πρόβλημα, το, ο ρόλος της αποθήκευσης της ενέργειας στο σύστημα της ενέργειας. Αλλά ο κύριος Γιώργος Χατζημαρκάκης ξεκίνησε με το δεύτερο πάνελ που το τίτλος του είναι οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας για τους τελικούς χρήστες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη της Επιτροπής. Στην ομιλία μου θα μιλήσω υπέρ ε, της αποθήκευσης και τελεία, χωρίς συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Παρότι εμείς είμαστε πάροχος ε, συγκεκριμένων συσσωρευτών, να σας ε, αναφέρω συντομία ποιοι είμαστε και τι ακριβώ κάνουμε. Αποστολή τη Τέσλα είναι να αλλάξει τον κόσμο, να συμβάλλει στην, ε, στο πέρασμα προς ε, μια εποχή βιώσιμης ενέργειας. Θέλουμε ουσιαστικά να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα στη φορά την παραγωγή ενέργειας και να βελτιώσουμε την κατάσταση για όλου. από κοινού βέβαια με την παραγωγή ε, εξαιρετικά όμορφων αυτοκινήτων και άλλων ε, προϊόντων. Να σας πω δύο λόγια για το τι ακριβώς ε, κάνουμε, τα προϊόντα μας που υπάρχουν ήδη στην αγορά και ήδη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και οι καταναλωτές πιο συγκεκριμένα ενεργούν και λειτουργούν. Εδώ έχετε το ζήτημα των τομέα των κατοικιών, βλέπετε εδώ στην αριστερή εικόνα Χιλιάδε τέτοιε εγκαταστάσει ε, κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή και τοποθετούνται στην Ευρώπη με φωτοβολταϊκά συστήματα που υπάρχουν δηλαδή ενσωματωμένα εκεί. Βλέπετε και το όραμά μας ε, ε, για την παραγωγή και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού που θα βοηθήσουν και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν αυτούς τους συσσωρευτές. Είναι κάτι το οποίο μας εμπνέει ιδιαίτερως σε εμπορικό επίπεδο. Εδώ βλέπετε μια κατάσταση που χτίζουμε στα Χαβάη αυτή τη στιγμή. Ένα ηλιακό σύστημα 13 μεγαλοβατόρων. Αυτό είναι ένα ε, σύστημα σε εμπορική κλίμακα, ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, αποθήκευση ενέργειας με στου ορεφτές, όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντε. Σημαντική προσπάθεια για την ε, ενίσχυση του δικτύου ή για ένα σύστημα μικροδικτύων όπως είναι αυτό ή με βάση την ανταπόκριση στη ζήτηση. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Αυτό είναι κάτι που ήδη υπάρχει στην αγορά. Δεν είναι ένα επιστημονικό μόνο εγχείρημα. Το βλέπουν και οι καταναλωτέ σε επίπεδο κατοικιών, αλλά και σε ε, βιομηχανικό επίπεδο, όπου οι επιχειρήσει προσπαθούν να ελέγξουν τι συμβαίνει ε, με βάση τη ζήτηση. Αυτό συμβαίνει ήδη σήμερα. Χωρί καμία άλλη στήριξη. Επομένω, βλέπουμε ότι και η αποθήκευση προσφέρει μεγάλη ικανότητα γιατί βλέπουμε ότι πλέον ε, παροπλίζονται παλαιότερες εγκαταστάσεις, ε, άνθρακα και ούτω καθεξής, αντί ε, να εγκαθιστούμε νέες μονάδες, βλέπουμε ότι η αποθήκευση ενέργειας έρχεται και υποκαθιστά τις προηγούμενες υποδομές με πολύ χαμηλότερο κόστος και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για τα κράτη-μέλη και την Ένωση του συνολό Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. καθώς αυξάνεται το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας και της αιωλικής. Ε, σαφώς ε, είναι κρίσιμη σημασία στη σταθεροποίηση του συστήματος, του δικτύου, ε, με την αποθήκευση ενέργειας πολλών διαφορετικών μορφών, κρίσιμη σημασία στοιχείο και θα μας επιτρέψει και να, καθώς θα μειώνεται το κόστος των ανανεώσιμων, να αυξήσουμε το μερίδιό τους στο ενεργειακό μας μείγμα. Και αυτή ήταν και η περιοριστική διάταξη μέχρι τώρα, ο περιορισμό που είχαμε μέχρι σήμερα. Για να σα δώσω μια εικόνα τη κλίμακα, οι συσσωρευτέ. Εμεί είμαστε γνωστοί ακριβώ για του συσσωρευτέ μα. Η τεχνολογία λοιπόν στι συσσωρευτέ δεν ε, είναι στάσιμη. Έχουμε πολύ σημαντικέ τεχνολογικέ εξελίξει. Ε, αυτή αφορά την ενεργειακή πυκνότητα, αλλά για να σα δώσω μια ιδέα ε, ενό στοιχείου σωρευτή, το οποίο δεν είναι στάσιμο, βελτιώνεται η τεχνολογία και αυτό οδηγεί και σε σημαντική ε, περικοπή του κόστους και γι' αυτό στο μέλλον θα έχουμε συσσωρευτές σε κάθε σπίτι. Η παγκόσμια αγορά τώρα για αυτά τα στοιχεία συσσωρευτή. Ε, ολοκληρώσαμε αυτό που αποκαλούμε Gigafactory. Μάλλον τώρα κατασκευάζεται ε, και θα κατασκευάζει ενεργειακά προϊόντα Τέσλα. Ουσιαστικά θα έχει την ίδια ικανότητα που είχαμε το 2014 για όλους τους τύπους. Ουσιαστικά δισεκατομμύρια λοιπόν δολαρίων και ευρώ στην αύξηση της κλίμακας, ούτως ώστε η χρήση αυτών των μπαταριών να είναι οικονομικά αποδοτικές και για τις ανανεώσιμες και για τις υπόλοιπες. Τώρα, οι στόχοι της ε, Ένωσης, πενταπλή. Ε, και η αποθήκευση τους ε, στηρίζει και τους πέντε στόχους. Δεν θέλω να τους αναφέρω όλους εξωδικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα αναφερθώ σε δύο μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει μεγάλο μερίδιο του πετρελαίου, του φυσικού ακόμα και του άνθρακα αυτή τη στιγμή στις ΕΕ. Ε, και η ενεργική ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό για μας ως ε, Ευρωπαίους, μας απασχολεί. Εδώ έχετε μία εκτίμηση από διάφορες ε, εκθέσεις για το υψηλότερο ποσοστό ικανότητας παραγωγής από τις ανανεώσιμες. Τι θα απαιτείται ως προς την αποθήκευση για να σταθεροποιήσουμε το δίκτυο μέχρι και το σημείο όπου το 100% της παραγωγής θα είναι από ανανεώσιμες. Ελπίζουμε αυτό να συμβεί ε, όσο ζούμε εμείς, αλλά εδώ σας δίνω μόνο ένα δείκτη. Γι' αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη Τέσλα, εμείς ηγούμαστε βέβαια αυτού του κλάδου στους συσσωρευτές, στη στατική αποθήκευση, αλλά και για, του, και για τις άλλες μορφές ε, αποθήκευσης ε, που έχουν αναφερθεί εδώ. Αυτό που χρειαζόμαστε, και το ακούσαμε και προηγουμένως, είναι να διασφαλίσουμε ότι οι οδηγίε θα επιτρέπουν την πρόσβαση ε, τη αποθήκευση ενέργεια στι επιμέρου αγορέ και δεν θα την παρεμποδίζουν με το να την ε, θέτουν σε στεγανά ε, ένα πεδίο που το, λέμε παραγωγή και ένα άλλο που το λέμε μεταφορά ενέργειας, γιατί αυτό ε, θα επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη του κλάδου. Ακόμα και αν δεν έχουμε ανανεώσιμε αποθήκευση με συσσωρευτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά για τη στήριξη του δικτύου όταν υπάρχουν αδυναμίες ε, και όταν έχουν ε, παροπληστεί, έχουν τεθεί εκτός λειτουργία σε μονάδες παραγωγής ενέργειας. Μπορεί λοιπόν η αποθήκευση να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση ε, σε σχέση με άλλες. Ακόμα και χωρί καμία λοιπόν αύξηση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, αν και εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ε, ε, αύξηση, παρόλα αυτά και πάλι έχει νόημα και λογική ε, να στραφούμε προς την αποθήκευση, γιατί τελικά το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο και για τον τελικό καταναλωτή. Δεν έχω πολύ χρόνο, προχωρώ λοιπόν. Με την αποθήκευση μπορούμε πλέον να περάσουμε σε έναν ε, τομέα ε, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε το κόστος της μεγάλης παραγωγής ε, και των υποδομών που κανένας δεν θέλει να αναλάβει το κόστος για αυτές και ουσιαστικά μπορούμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά στο δίκτυο και να το σταθεροποιήσουμε και να αρχίσουμε τη λειτουργία του πολύ πιο γρήγορα και οικονομικά. Θέλουμε λοιπόν πλέον να περάσουμε στην ε, μεταφορά ε, όχι ηλεκτρονίων αλλά δεδομένων και ενέργειας που είναι πολύ πιο σημαντικό για εμάς. Κλείνοντας, τελευταία διαφάνεια, για τον κατανολωτή, τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, τι αλλάζει, αλλάζουν οι συμπεριφορές ε, αλλάζει η νοοτροπία όταν κατανοεί ο καταναλωτής ότι μπορεί ο ίδιος να χειρίζεται και τις πληροφορίες και τις, ε, έχει τις επιλογές για το πώς θα αξιοποιεί την ενέργεια και πλέον και ο ίδιος ο θα μπορεί να ε, ε, διαχειρίζεται την ενέργειά του και να μην εξαρτάται από μεγάλες επιχειρήσεις και έχουμε ενέργεια που θα χορηγείται από έναν ε, ενεργειακό τοίχο, wall, Και αυτό θα επιτρέπει στον καθένα μας, όποτε θέλουμε, να έχουμε πρόσβαση στην ενέργεια και να ξέρουμε τι θα πληρώνουμε. Στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε ευφυείς μετρητές και οι χρεώσει θα είναι πιο αυξημένε όταν είναι και μεγαλύτερη ζήτηση και ο κάτι που στο ιδιοκτήτη του σπιτιού θα μπορεί να προγραμματίζει αναλόγως και το συσσωρευτή και να χρησιμοποιεί έτσι ενέργεια με χαμηλότερο κόστο. Συνολικά λοιπόν ήδη είναι συμφέρουσα λύση η αποθήκευση, προχωρούμε γρήγορα, χρειαζόμαστε στήριξη ούτω ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί σε ό,τι αφορά την αποθήκευση. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να αρχίσει συζήτηση. Ρουμπιχ Κόχλιτσα και είναι οι και έπονται συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ε, Κύριε Ρουμπιχ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά ε, για τη ματιά που μας αφήσατε να ρίξουμε σε μεγάλο βάθος στην αγορά ή στις αγορές της αποθηκεύσης είναι τεράστια ευκαιρία για τις ΑΠΕ για να διαθέτουμε και τις ανανεώσιμες. Η πρώτη αρχή είναι ότι χρειαζόμαστε τα δίκτυα, τις υποδομές, να τα επεκτείνουμε έτσι ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να μπορεί να μεταφέρεται. Ε, και εκείνη που μπορεί να αποθηκεύεται, αλλά και οι άλλες ενεργειακές μορφές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό που θα με ενδιαφέρει να ακούσω από την Τέσλα είναι η διάρκεια ζωή ενό συσσωρευτή και η χρήση εξαρτάται ε, εάν είμαστε ε, σε πόλη που έχει πολλά φανάρια και σταματάς από φανάρι σε φανάρι, όπως είναι το Στρασβούργο, που ε, ε, συνειδητά διαρκούν ε, ώρες τα κόκκινα για να κυκλοφορούν τα τραμ και δημόσιες συγκοινωνίες εστικές. Η Τέσλα το έχει σκεφτεί αυτό, μήπως να μπορεί να δημιουργήσει πράσινα κύματα με τους νέους αλγορίθμους έτσι ώστε στις ευφυείς πόλεις να υπάρχει απρόσκοπτη και πιο ομαλή ε, κυκλοφορία από το σημείο Α ή από το Β και αυτό δεν εξαρτάται από το αυτοκίνητο μόνο ή από το συσσωρευτή αλλά από τις υποδομές στις ευφυείς πόλεις äh, που δεν ε, Ε, πρέπει να φρενάρουν τα αυτοκίνητα γιατί από εκεί έχουμε όλο αυτό το νέφος, ε, όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια γιατί τρίβονται τα ελαστικά, το καουτσούκ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ε, βασικά και στη ΣΤΟΑ που ξέρετε ότι είναι η επιστημονική μας επιτροπή στο Κοινοβούλιο, Scientific and Technology Options Assessment είναι η ΣΤΟΑ, εξαρτάται πάρα πολύ από τις στάσεις και τα φρεναρίσματα. Το ίδιο και με το σιδηρόδρομο. Ε, είναι πιο αποτελεσματικός και πιο αποδοτικός ε, όσο το τρένο βρίσκεται στις ράγες και κυκλοφορεί και δεν πρέπει να φρενάρει, να σταματάει, να ξαναρχίζει και δεν συμμαζεύεται. Εκεί χρειαζόμαστε κάποιους αισθητήρε και αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για μένα, όχι το ίδιο το αυτοκίνητο, αυτή είναι η παλιά νοοτροπία. Η νέα νοοτροπία είναι αυτή. Πώς θα είναι η ροή έτσι ε, και η κυκλοφορία μάλλον πιο ρευστή χωρίς ε, στάσεις. Ευχαριστώ ε, από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευρώπα 40% Κύριος Γκίρεκ. Ευχαριστώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ενέργεια που να μπορεί να αποθηκεύεται και να τη χρησιμοποιούμε και για θέρμανση και για ψήξη. Ε, έχουμε εδώ λοιπόν πολύ χρήσιμες ε, εφαρμογές σε αυτό το τομέα, διότι τα δίκτυα και ο ηλεκτρισμός είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιλύσουμε σε μακρο, σε μακρο κλίμακα. Ενώ ε, όταν πρόκειται για θερμότητα είναι διαφορετικό είδο ενέργειας και θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι ενδεχόμενες προοπτικές χρήσης αυτών των μεθόδων για τη θέρμανση. Ποιο από αυτά τα συστήματα έχει το περισσότερο και καλύτερο μάλλον δυναμικό ιδιαίτερα από την άποψη της μετατροπής της ενέργειας διότι εάν η αλυσίδα μετατροπής είναι ε, μακρά ε, δεν θα έχουμε πολλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι... Greens. Ευχαριστώ που έπανε ο ο κ. από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με, τα με όσους είπατε ότι ε, ίσως δεν πρέπει να αποφασίσουμε τώρα ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε με όλες αυτές τις δυνατότητες, αλλά ότι ε, πρέπει να υπάρχουν, να δίνεται δυνατότητες για πολλά πράγματα εδώ. Είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια με το πιο αποτελεσματικό τρόπο στο μέλλον, αλλά πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον να δούμε εταιρείε που χρησιμοποιούν την αποθήκευση σε ένα μεσαίο επίπεδο μεγέθους. Το, όταν είναι, το αγοράζουν όταν είναι πολύ φθηνό και το πολλούν όταν οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι υψηλότερες. Και νομίζω πως η αγορά θα πρέπει να υπάρχει ήδη, θα έπρεπε να υπάρχει ήδη θα έπρεπε να υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής, γιατί υπάρχουν, όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σήμερα στις αγορές ενέργειας. Οπότε θα πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα για να αγοράσει κανείς πολύ φθηνό ηλεκτρισμό και να το πουλήσει όταν ε, αλλάζει η κατάσταση. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα είναι, είδα κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον είχαμε μια συζήτηση για το χάλιβα στην Ευρώπη. Η χαλιβουργία χρησιμοποιεί πάρα πολύ άνθρακα. Πολλές εκπομπές έχει και καταστρέφει το κλίμα. Αλλά η Σουηδική Χαλιβουργία είχε αυτήν την ιδέα τώρα αυτό που θέλουν είναι να αναπτύξουν τη χρήση του υδρογόνου για να κατασκευάζουν το χάλιβα αντί για τον άνθρακα. Πιστεύετε πως είναι μια λύση αυτή που θα καταστεί δυνατή στο μέλλον. Γιατί εάν αυτό είναι κάτι που γίνεται θα μπορούσε να απορροφήσει τεράστιους ε, όγκους ευθυνού ηλεκτρισμού και να παίξει ένα πολύ μεγάλο, να, να αποτελέσει μάλλον ένα μεγάλο τμήμα της λύσης. Να παράγουμε ευθυνή, δηλαδή ηλιακή και ολική ενέργεια, να τη δίνουμε στη Γαλλιβουργία αντί για τον άνθρακα. Thank Σας ευχαριστώ. Α, όχι, γκουε. Όχι. Ε, ναι. Εγώ είμαι ε, επιχειρηματία. Και έχω τρία, τρεις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με 4,1 κιλοβάτ ανώτατο, ανώτατη παραγωγή και δύο, οι άλλες 2,7. Οι δύο ε, παρέχουν στο πλέγμα βέβαια οι εταιρείε δεν, με δεν με πληρώνουν πολύ περισσότερο. Το τρίτο μου, ε, η τρίτη μου μονάδα χρησιμοποιεί Ε, ε, χρησιμοποιεί συσσωρευτές γιατί είναι στο εξοχική μου κατοικία ε, και εκεί είναι καλύτερη κατάσταση. Πριν από πέντε χρόνια ένας διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε το 2020 το 1% της ενέργειας στην οικονομία του υδρογόνου. Έκτοτε δεν έχω ακούσει ούτε μια λέξη σε σχέση με την εφαρμογή όλων αυτών στην Τσεχία. Στο στην Τσεχία, στο Νεράτοβιτσε, έχουμε μία μονάδα υδρογόνου, έχουμε τα λεωφορεία που χρησιμοποιούν οι Είναι λογικό, είναι καθαρό, δεν χρειάζεται καμιά μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, είναι σπουδαίο, είναι μια πολύ κομψή λύση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, γιατί είναι τόσο μικρή η χρήση. είναι πολύ ελκυστικό. Τόσο μικρή μονάδα που έχω εγώ, δηλαδή 4 κιλοβάτα, αν έχει κάποιο πλεόνασμα, αν μπορούσε και να αποθηκεύσει την ενέργεια, δεν χρειάζονται μεγάλες μπαταρίες. Γιατί οι σημερινές μπαταρίες έχουν και πολύ μικρό κύκλο ζωής. Χαλάνε γρήγορα, ειδικά αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτή την ενέργεια. Αυτά που συζητάμε λοιπόν είναι πολύ πρακτικά. Είναι πρακτική λύση και για μένα και πραγματικά προσβλέπω στην ημέρα όπου θα μπορούσα να έχω ε, μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια μονάδα στο σπίτι μου, να μπορώ να το χρησιμοποιώ γιατί εγώ ε, είμαι φίλος της τεχνολογίας και αυτό που λέμε εδώ θα πρέπει να εφαρμοστώ στην πράξη, να δείξουμε δηλαδή στον κόσμο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο λόγια, ε, μιλάει για πράγματα που έχουν καθημερινή χρήση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο ε, Σάβεγκα. για αυτή την ε, σε βάθος παρουσίαση αυτών των σημαντικών ζητημάτων όπως είναι η αποθήκευση. Κατανοούμε βεβαίω ότι είναι κρίσιμο ζήτημα από ορισμένε πτυχές αποθήκευση, είναι αναπόφευκτο μάλιστα. Είπατε ότι η αποθήκευση μπορεί να διαναμηθεί σε πολλές πλευρές ε, και από την πλευρά του παρόχου, ε, του ενδιαμέσου και του καταναλωτή. Αυτό είναι διαφορετικό για παράδειγμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν έχουμε αρκετού τέτοιου σταθμού ε, αποθήκευση και αυτό είναι πρόβλημα και τροφοπαίδευση στην εξέλιξή του. Από την άλλη, έχουμε, λέμε ότι και αυτά τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση σε μεγάλη κλίμακα. Είναι πιο εγωιστικό το δικό μου ερώτημα. Υποκειμενικό. Ε, εργάζομαι στην έκθεση του κυρίου Γκίρεκ για την ε, ψήξη και θέρμανση και αναφέρατε ότι και στη θέρμανση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πλευράς καταναλωτή να υπάρξει δηλαδή και κάποιο είδους αποθήκευση. Μπορείτε να μας ε, το αναλύσετε αυτό λίγο. Τι είδου ε, προβλήματα εσεί ε, εντοπίζετε, Υπάρχουν νομικά προσκόμματα, οικονομικά. Και αυτό που παρατηρώ εγώ, έχοντα δει τα ζητήματα θέρμανση και ψήξη, το πιο σημαντικό είναι η παροχή κινήτρων. Η ενθάρρυνση του τελικού καταναλωτή. Πώ θα παροτρύνουμε λοιπόν τον καταναλωτή να συμμετάσχει σε τέτοιου είδου ε, προσπάθειε. Δεν ξέρω, όποιο θέλει να μου απαντήσει. Να μου δώσει ορισμένα προσφέρα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος ε, του καταλόγου μιλητών. Να προσθέσω από πλευρά μου ένα ερώτημα προς τον Γιώργο Χατζημαρκάκη. Στις αρχές ε, του τρέχοντος αιώνα, πριν από 15 χρόνια δηλαδή, είχαμε πολύ περισσότερες, μεγαλύτερες προσδοκίες από την οικονομία του υδρογόνου. Και ο καθηγητής ε, Ρίφκιν από τις ΗΠΑ έφτασε στην Ευρώπη και μας είπε ότι το 2010, όχι πιο μετά, θα μπορούσε κανείς να αγοράσει έναν συσσωρευτή υδρογόνου σε οποιοδήποτε κατάστημα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κίνα, οπουδήποτε. Κάτι συνέβη. Δεν ξέρω πότε. Ίσως μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε περαιτέρω. Αλλά μπορείτε να μας πείτε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από τις προσδοκίες που είχαμε πριν από 15 χρόνια σε σχέση από την οικονομία του υδρογόνου και από το υδρογόνο ως ε, μορφή αποθήκευσης. Στην Ισλανδία υπάρχει δυνατότητα λόγω θερμικών ε, πηγών. Αλλά πώς όλα αυτά συνδέονται με το σήμερα και τι θα γίνει και στο μέλλον. Πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω. Και ένα ερώτημα προς όλους τους εξαιρετικούς ε, ομιλητές. Μπορείτε να μας δώσετε μία ημερομηνία, σύν πέντε χρόνια όπου θα μπορούσαμε να σταματήσουμε το backup φυσικού αερίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, μονάδες φυσικού αερίου ως ε, εφεδρεία ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε μεγάλη κλίμακα τώρα λέω. Αυτά τα δύο ερωτήματα έχω. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολα, αλλά Ας ξεκινήσουμε από αυτά, ίσως με την ίδια σειρά, αν ε, θέλετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ για το πολύ εύκολο αυτό το τελευταίο ερώτημα. Μισό λεπτό να βγάλω τη γυάλινη σφαίρα μου κρυστάλλινη. Ε, θα ήθελα να πω για το όσο είπε ο κύριο Ρούμπικ ότι δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Πρέπει να έχουμε το συνολικό σύστημα στο οποίο θα ενταχθεί κάποια τεχνολογία. Τώρα πώ θα γίνει αυτό στην πράξη και λεπτομερώς δεν το ξέρω, λοιπόν, πρέπει να τα δούμε για τα δύο που κοινού. Και το σύστημα και τι τεχνολογίε εντό του συστήματο. Ο κύριο Γκίρεκ ρώτησε για τη θέρμανση και ψήξη και το ίδιο ακούσαμε και στη συνέχεια. από πολλές μελέτες, αλλά και ο συνάδελφος θα επεκταθεί στη συνέχεια, ότι η αποθήκευση θέρμανσης είναι πιο οικονομική και η προσθέμενη αξία είναι ότι μπορούμε να πάμε από τον έναν φορέα, από την ηλεκτρική ενέργεια, τη μία μορφή στην άλλη, από την ηλεκτρική ενέργεια, στην ε, θέρμανση, ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις μεταφορές, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε σωρευτές, στα οχήματα, και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι ήδη. Ένα από τα μέλη μας λοιπόν, μια Ιρλανδική επιχείρηση, ήδη σήμερα παρέχει τη δυνατότητα εφιούς ε, θερμικής ε, αποθήκευσης, δηλαδή μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει ε, ενέργεια για να χρησιμοποιήσει ως θέρμανση. Και αυτή η θέρμανση μέσω του boiler είναι, ε, ελέγχεται από τους DSOs ή DSOs και τίθεται σε λειτουργία όταν έχουμε πολύ αέρα. Όταν δηλαδή οι τιμές ενέργεια είναι πολύ αρνητικές ή έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας, τότε ξαναμπαίνουν. Τώρα, γιατί δεν έχουμε παραπάνω τέτοιες τεχνολογίες. Πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να πουλήσουμε αυτή την ευελιξία στην αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν aggregator που θα τα συγκεντρώσει όλα αυτά και θα τα πουλάει και η ανταπόκριση από πλευρά ζήτηση δεν παρουσιάζει την ίδια κατάσταση στην Ευρώπη με τι ΗΠΑ. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ε, εξετάσουμε το σχεδιασμό τη αγορά για να μπορέσουμε να συγκερέσουμε τα επιμέρους στοιχεία και την, ε, από πλευρά ζήτηση και προσφοράς σε μία ενιαία αγορά. Για να απαντήσω τώρα ε, για τους διαμεσολαβητές, το arbitrage όπως ε, ρώτησε ο κύριος Έριξον, είναι κάτι το οποίο ε, είναι θετικό. Δηλαδή, οι τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια διατρίζουν ε, την πραγματική αγορά. Δηλαδή, αν έχουμε έλλειψη ευελιξίας ή έλλειψη προσφοράς, ε, αυξάνονται τιμές, υπερβολική προσφορά χαμηλώνουν οι τιμές και ούτω καθεξής. Από πλευρά σχεδιασμού της αγοράς, λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτή η τιμολόγηση να διέπει όλο το σύστημα και να φτάνει μέχρι τον καταναλωτή. Αλλά τελικά έχουμε και κοινωνικό ζήτημα θέλουμε να εκθέσουμε τον καταναλωτή σε έναν σενάριο να πληρώνει 2, 3, 4 χιλιάδες ε, ευρώ την κιλοβατόρα, ακόμα και αν είναι για ένα λεπτό, για πέντε λεπτά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πού βάζουμε το όριο. Πρέπει να είναι μόνο για τους ε, καταναλωτές, ε, του βιομηχανικού, και μετά στη λιανική υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Αυτό είναι θέμα πολιτική απόφαση. Όμω, ε, το arbitrage είναι όντω ένας από τους τρόπους που να ακολουθήσουμε για την αποθήκευση. Και ε, ο εξοπλισμό αποθήκευση πρέπει να αξιοποιήσει όλους, ε, όλες τις και για την εξορρόπηση του συστήματος και για την διαμεσολάβηση αυτή του arbitrage και για να φτάσει στο τελευταίο. Θέλετε να σας δώσω μια χρονική στιγμή πρόβλεψη, δηλαδή για το πότε δεν θα χρειαζόμαστε εφεδρείες φυσικού δεδομένων των τεράστιων ε, αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια αυτή τη στιγμή στην ε, Ευρώπη, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα το ζήσουμε εμείς τουλάχιστον. Μάλιστα. Για να απαντήσω ε, και πάλι για τη θέρμανση, λέει ο κ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξή. Δεν λέμε ότι έχουμε ένα σύστημα θέρμανσης. Βεβαίως η θέρμανση είναι πάρα πολύ ε, αποκεντρωμένο και από την άλλη ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον, αυτά τα δύο θα μπορούσαν να συγχωνευτούν ουσιαστικά και όλο περισσότερο να παράγουμε θερμότητα από ηλεκτρική ενέργεια με ε, ανανεώσιμες. ανανεώσιμες ε, και τα φωτοβολταϊκά και η ελληνική ενέργεια σε πρώτο λόγο παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το θέμα τώρα το ρεύμα, πώς μπορούμε μέσα σε ένα νοικοκυριό, σε ένα σπίτι να το μετατρέψουμε με τρόπο αποτελεσματικό. Και έχουμε μια τεχνολογία που είναι ε, η αντλία θέρμασης, η οποία δεν μπορεί όμως να εγκατασταθεί σε κάθε σπίτι. Άρα, πρόθεσμα θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κατασκευές κατοικίες για να μπορούμε να έχουμε τέτοιες αντλίες για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε πραγματικά τις ανανεώσιμες να μπαίνουν σε αυτό το σύστημα. Ε, ένα αριθμητικό στοιχείο μόνο. Στη Γερμανία έχουμε 600 τεραβατόρες για ε, τα νοικοκυριά. Αν το κάνουμε αυτές τις αντλίες θα μειωθεί στο 1 τρίτο αυτό. Μάλλον ένα τρίτο επιπλέον, συγγνώμη. Δεν είναι καμία τεράστια ε, πρόοδο, καμία τεράστιο άλμα αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το καταλάβουμε και τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Δεύτερη ερώτηση, επόμενη, για το υδρογόνο. Ρώτησε κάποιο τι γίνεται με το υδρογόνο στην ε, Χαλιβουργία, ο κύριο Έριξον. Ναι, το μελετήσαμε αυτό. Ποτέ βέβαια δεν δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη. Μαζί με τη Siemens ε, το μελετήσαμε πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ως καύσιμο το υδρογόνο σε μια ε, χαλιβουργία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα και η τεχνολογία. Αλλά πρώτα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ήδη από σήμερα χρειαζόμαστε πολύ ε, υδρογόνο στις χημικές βιομηχανίες. Για να κάνεις αμμονία χρειάζεσαι υδρογόνο. Ή Ακόμα και στα δηληστήρια χρειάζεται πάρα πολύ υδρογόνο. Πριν ανοίξει νέα αγορά, η χαλιβουργία, καλό θα ήταν να καλύψουμε τις αγορές που ήδη υπάρχουν, διότι ε, δεν χρειάζεται μεγάλη αναδιάρθρωση σε αυτό. Ε, από την άλλη, σε πολύ μακρόπνοη έτσι, κατάσταση, ε, χρειάζεται υδρογόνο ενδεχομένω και στη χαλιβουργία, αλλά δεν είναι του παρόντος ούτε του αύριο. Κάτι άλλο που ρωτήσατε, γιατί δεν έχουμε ήδη από τώρα την οικονομία του υδρογόνου. Και ήταν κάτι παραπλανητικό στη δεκαετία του 90. Κυκλοφόρησε αυτή η ιδέα ότι τα στοιχεία ισορρευτές ε, καυσίμου θα ήταν πολύ φθηνά. Ε, θα ήταν τόσο φθηνά όσο ο κινητήρα σήμερα. Ε, 50 με 100 ευρώ ε, το κιλοβάτ, αλλά αυτή ήταν παραπλανητική ιδέα. Βεβαίω, αν είχε συμβεί, θα άλλαζε και η αγορά και η νοοτροπία και η κατασκευή των αυτοκινήτων. Και τέλος, για την τελευταία ερώτηση, νομίζω το 2050 ακόμα θα έχουμε αποθέματα και εφεδρείες φυσικού αέριου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε και ένα δεύτερο μοντέλο. Το ένα είναι για τον ηλεκτρολίτη, πώς παράγει υδρογόνο και το χρησιμοποιεί. Και έχουμε την Κατερίνα Μπόμελμποκ από, το, από που θα σα εξηγήσει πώς λειτουργούν αυτά. Και έχουμε για στατική αποθήκευση για την ε, θέρμανση. Και ε, έχουμε από τις ενεργειακές λύσεις... Ε, ε, για να απαντήσω στον κύριο Έριξον, καλύφθηκε η απάντηση από τον καθηγητή Χάμαχερ και ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Λέει ότι είναι μακράς πνοής αυτή η όγκη του υδρογόνου. Δεν είμαι τόσο βεβαίω. Ε, όταν έχουμε υπερβολική ενέργεια που δεν τη χρησιμοποιούμε, θα μπορούσαμε, ας πούμε, δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα να κινούμε με υδρογόνο. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά τους μεγάλους όγκους βεβαίως ε, θα τους χρησιμοποιήσουμε στα δηληστήρια, Φερρυπίν. Εκεί, χωρίς εκπομπές ρήπων, υπάρχει αντικατάσταση, δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, ε, καυσίμων, ε, που τελικά στο μείγμα και στο αποτύπωμα άνθρακα είναι εξαιρετικό. Ποιος έφυγε? Α, ο Παύλος Ρουμπιχή δεν έφυγε, προεδρεύει κιόλας. Για τη δική σου ερώτηση, για τις ευφυείς πόλεις, εγώ θα το πήγαινα ακόμα παραπέρα. Ας πούμε τι γίνεται με ε, τους ευφυείς διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Τώρα μιλάμε ε, ε, πώς θα ξεφύγουμε από το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει οι εμπορευματικές μεταφορές ε, γίνονται όλο και περισσότερο από μεγάλα βαριά φορτηγά που καίνε ντίζελ και δεν πάνε στο σιδηρόδρομο. Άρα ε, αυτοί οι διαδρομοί πολύ απλά μπορούν να δημιουργηθούν με όπου να έχουμε πραγματήρια καυσίμων υδρογόνου με πρότυπα. Έχουμε διαφορετικές ε, μορφές τυποποίησης της αντλίας για το υδρογόνο. Ε, εάν αυτό το τυποποιήσουμε, μπορεί κάποιος να πάει από τη Σικελία στην Κοπενχάγη, ξέρω εγώ, ε, με βαρύ φορτηγό και να ε, γεμίζει το ντεπόζιτο με υδρογόνο. Κάτι που είπα στην παρουσίαση επίσης, με τα στοιχεία αυτά καυσίμου μου σωρευτές, η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μπορεί να εξοικονομηθεί κατά 60% που είναι αρκετά μεγάλο. Ο κύριος Κόχλιτσε τα ξέρει πολύ καλά, είναι μέγας ε, ε, υποστηρικτής ε, και πέρμαχος αυτής της τεχνολογίας και αυτό ισχύει και για μεγάλες και για μικρές εφαρμογές. Εγώ ως πρώην Ευρωβουλευτής να σας πω το εξή. Ήρθα στο Κοινοβούλιο το 2004 και είχαμε τότε αυτή τη μόδα και τη μανία με τα βιοκαύσιμα. Χαμός γινότανε. Δεν μπορούσες να ξεφύγεις από συζήτηση για τα βιοκαύσιμα. Από πουθενά. Ε, κάναμε και πολλή νομοθεσία, θυμάστε. Και μετά από δύο-τρία χρόνια σταμάτησαν τα πάντα. Κιχ δεν ακουγότανε. Αυτές είναι μόδες που είναι αρκετά επικίνδυνες. Διότι η πολιτική και η κοινή γνώμη και οι πάντες παραπλανούνται. Τώρα δεν θα διαπλεκτιστούμε, αλλά έχω την ε, εντύπωση ότι η μόδα αυτή και η μανία για τους ισορρευτές μου θυμίζει κάποια στοιχεία εκείνης της ε, συζήτησης. Είμαι βέβαιος ότι χρειαζόμαστε μπαταρίες οπωσδήποτε στο μείγμα, αλλά μην μας πιάνει τρέλα γιατί αυτό θα ε, είναι εις βάρος της ανάπτυξης ε, του ηλεκτρισμού γιατί θα φτάσουμε στα όρια μας και ο κόσμος θα απογοητευτεί και θα γυρίσει την πλάτη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κύριε Σαουντάργα, σε ευχαριστώ πολύ. Ρωτήσατε γιατί κάποιες τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Λουξεμβούργο, το νέο κτίριο Κόνρατ Αντεναόερ του Κοινοβουλίου, ε, στο διαγωνισμό, στην αρχή είχε συσσωρευτές με μηδενικές εκπομπές και Μπαταρίε ή λιγότερε εκπομπέ εμπάσει περιπτώσει. Έτσι, το έλεγε ο διαγωνισμό, πάση περιπτώσει. Έτσι, το έλεγε ο διαγωνισμός, η λιγοτερε εκπομπες εν παση περιπτωσει ετσι το ελεγε ο διαγωνισμο ήρθαν οι προσφορές και οι τιμές και σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όχι ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, αποφασίστηκε ότι είναι πανάκριβο, όχι χαίρεται. Βλέπετε, ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν συζητήθηκε αυτό στις επιτροπές, αλλά σε χαμηλό επίπεδο διοίκηση ε, το απέρριψαν επειδή είναι πολύ ακριβό. Μα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακριβό γιατί είναι στα σπάραγανα αυτή η βιομηχανία. Εάν δεν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας. Δυστυχώς ε, χρειάστηκε να αποχωρήσει ο Γέρζε που έκανε τη βασική ερώτηση. Τι λάθος έκανε, τι σωστό έκανε ο κύριος Ρίφκιν στην οικονομία του υδρογόνου. Ε, ε, ε ειδικοί, ε, οι υποστηρικτές και οι οπαδοί ε, αυτού του κλάδου θεωρούν ότι ο κύριος Ρίφκινγκ δεν τα πήγε καλά και δεν έκανε ε, καλή δουλειά. Γιατί, γιατί φούσκωσε πάρα πολύ τις ελπίδες και χρειάστηκε να το πουλήσουμε πάρα πολύ, να τάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Το κάνεις αυτό, το κάνεις δύο-τρεις φορές και μετά ε, χάνεις την αξιοπιστία σου. χάσαμε λοιπόν με πολλές ευκαιρίες και πολλή αξιοπιστία. Είναι γεγονός. Και κατά τα άλλα ο κύριος Ρίφκινγκ δεν είναι πολύ γνωστό ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε για το υδρογόνο. Ίσως στην Καλιφόρνια, στην Ευρώπη είναι πιο γνωστό για το υδρογόνο. Και τώρα έχει έρθει ο καιρό και απαντώ εδώ στον Μπούζεκ μετά το COP21. Θα θυμάστε τι συζητήσει αυτέ που είχαμε αν υπάρχει υπερθέρμανση, όχι, χρόνια ολόκληρα. Τώρα δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι ε, η παγκόσμια κοινότητα δεσμεύεται προς την κατεύθυνση αυτή. Τελεία και παύλα. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα φτάσουμε εκεί. Η Greenpeace Στη τελευταία έκθεση που ονομάζεται η ενεργειακή επανάσταση εντός ε, ε, εισαγωγικών μιλάνε για το υδρογόνο σε 155 σελίδες 600 τόσες φορές. Αν θέλουμε να πάμε σε μηδενικές εκπομπές δεν είναι πάρα πολλές λύσεις. Τεχνικά είναι αυτή η εξή μία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα τελευταία πέντε λεπτά ανήκουν στον κύριο Χίλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για να δω αν τα έχω σημειώσει όλα. Έχουν ήδη απαντηθεί πολλά ερωτήματα. Το... Είναι καλό λοιπόν από αυτήν την άποψη να μιλάει κανεί τελευταίο. Σε ό,τι αφορά τι ευφυεί πόλει, υπάρχει η τεχνολογία, υφίσταται για την αυτόνομη οδήγηση. Πρέπει αρκεί να μπείτε σε ένα όχημα Τέσλα, να το δοκιμάσετε, να το δείτε κι εσεί ε, στην πράξη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία, δεν υπάρχει ακόμα ε, το κανονιστικό πλαίσιο που θα το επιτρέψει. Έχουμε πολλέ συζητήσει με την και Διεύθυνση Μεταφορών και άλλου ε, φορεί ε, στι Βρυξέλλε που θα μας επιτρέψει να απελευθερώσουμε και το οδικό σύστημα στην Ευρώπη. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς θα απομακρυνθούμε από τον άνθρακα στις μεταφορές, θα απεξαρτηθούμε και αν δείτε τις πόλεις μας, είναι τρομερά τα πράγματα. Δεν είμαστε στην Κίνα, είμαστε στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι και πάλι είναι επικίνδυνα τα πράγματα σε ό,τι φορά την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Αν δείτε για παράδειγμα την Ισπανία. Επομένω πρέπει να περάσουμε σε απεξάρτηση από τον άνθρακα στι μεταφορέ. Είτε πάμε στα ηλεκτρονικά οχήματα, αυτό είναι η καλύτερη επιλογή, είτε σε κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα, πρέπει πραγματικά να το εφαρμόσουμε σύντομα. Να βρούμε λύση. Για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ε, υπάρχουν ήδη αυτοί οι aggregators και τα επιχειρηματικά μοντέλα επίση διαμορφώνονται. Έχουμε στου ορευτέ. Ε, που ήδη εγκαθίστανται και αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και επιτρέπουν στους aggregators να εξοικονομούν, ε, μάλλον να βγάζουν χρήματα, να έχουν κέρδη και οι καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα. Αυτό δεν είναι από εκεί μας φαντασίες μας, υπάρχει ήδη σήμερα. Το μόνο που ζητούμε λοιπόν είναι να άρετε τυχόν εμπόδια για την εμπορική εξέλιξη μιας πραγματικής λύσης για τα ενεργειακά προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Σε διαφορετικό βαθμό στα επιμέρους κρατημέλη. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν είναι πολύ θετικό προς τον κύριο Κόλτσεκ. Εγώ χρησιμοποιώ το δικό μου φωτοβολταϊκό σύστημα για να φορτίσω το αυτοκίνητό μου. Αν δεν έχετε ηλεκτρικό όχημα, μπορώ να σας βοηθήσω κάποια στιγμή αν θέλετε. Αλλά μπορείτε να φορτίσετε το όχημα του ε, γειτονά σας και μπορείτε να βγάλετε και κανένα φράγκο. Υπάρχουν όμως ε, πολλοί τρόποι και πολλοί λόγοι. Ε, η αποθήκευση ενέργειας είναι τη σημασία ε, και βρίσκεται στο πυρήνα των όσων πρέπει να κάνουμε για το ενεργειακό μας ε, δίκτυο και ο σχεδιασμός αγοράς ε, μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα στους καταναλωτές και να δώσει σε όλους εμάς ω ιδιοκτήτες σπιτιών και, και, και ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και κατανόηση τη σημερινή κατάσταση. πολύ. Ήταν πολύ αποδοτική και αποτελεσματική η ακρόαση. Φορτίσαμε τις μπαταρίες μας για τις νέες δραστηριότητε αυτές. Μάθαμε πολλά πράγματα για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και αισθανόμαστε και ευθύνη τώρα εμείς να αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη αγορά γιατί θα βοηθήσει ε, όχι μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι παγκόσμιο το θέμα και το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις και όλα τα μέλη που παρέμειναν για την ενεργή του συμμετοχή στη συζήτηση και τους φίλους μας από την Επιτροπή και όλους τους παρόντες ε, και όσους μας ακούνε. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση 23 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι και 24 Μαΐου 9 με 12.30. Θα τα πούμε τότε. Ε, καλό σας ε, απόγευμα και ό,τι επιθυμείτε. Ε, και μπορείτε να δοκιμάσετε και το ποδήλατο, λέει ο κύριος Χατζημαρκάκης, αν θέλετε.